Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και είπατε εκπρόσωπα. Έχω λάβει έξι σχέδια ψηφίσματος από τις πολιτικές ομάδες. Θα ψηφίσουμε σε λίγο από τις 11.30 και μετά. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα και να ενημερώσω ότι ο Πρόεδρος έλαβε από το ΕΛΚ και το ECR Έτοιμα για να διορίσει τον κύριο Πασκάλα Ριμό ε,